proceeds with... Και τώρα η Επιτροπή Απασχόλησης ε, θα συνεχίσει στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης που αφορά την ε, τροποποίηση του κατεξουσιοδότηση ε, κανονισμού σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την Επιτροπή μας Θέλω να ελπίζω ότι υπάρχει κάποιος εδώ από την Κομισιόν, η κυρία Σούκοβα από την Επιτροπή από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, που ε, έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας πάνω σε, αυτή, ε, σε αυτό το θέμα. Είστε έτοιμοι να λάβετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρίσκομαι εδώ για να σας παρουσιάσω την πρώτη τροποποίηση σχετικά με τον κατεξουσιοδότηση κανονισμού που υιοθετήθηκε χθες από το Κολέγιο των Επιτρόπων στις 9 Ιουλίου και σύμφωνα με αυτό θα θέλαμε ε, να ορίσουμε την, ε, τον καταξουσιοδότηση κανονισμού και τον καθορισμό των τυποποιημένων ε, κλιμακών μοναδιού κόστος και των καταποκοπή ποσών για την επιστροφή των δαπανών των κρατών μελών από την Επιτροπή. Όπως αναφέρθηκε, αυτό υιοθετήθηκε πέρσι τον Ιούλιο και τέθηκε σε ισχύ στις 18 Δεκεμβρίου του 2017, ύστερα από την μη ένσταση του Συμβουλίου όσον αφορά το σημείο 41 ε, ε, θα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε από απλοποιημένες διαδικασίες ε, διότι η Επιτροπή θέλει μια απλοποιημένη διαδικασία καθώς επίσης και τον περιορισμό των ελέγχων, την απλοποίηση των ελέγχων διότι έτσι επιτρέπεται να επικεντρωθούμε περισσότερο στα αποτελέσματα από τις τους ελέγχους ε, ο καθορισμός των τυποποιημένων κλιματικών μονάδων κόστος μπορεί να, εφαρμοστεί ε, σε δημόσια έργα διότι αυτές οι εναλλακτικέ εφαρμόζονται σε αιτήματα τα οποία έχουν στείλει τα κράτη-μέλη στην Κομισιόν και δεν ταιριάζουν αναγκαία ε, στις, στα αιτήματα των αρχών. Αυτό επιτρέπει στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις δικές τους ε, πρακτικές και και ο κατεξουσιοδότης κανονισμός επιτρέπει ε, τη συμφωνία με τα κράτη-μέλη τα οποία, οποία είναι, συμμετέχουν σε αυτό τον κανονισμό και να προσαρμοστούν αυτόματα με το πέρας του χρόνου χωρίς ε, να υπάρχει ανάγκη επιβεβαίωσης ε, των αλλαγών. Μέχρι στιγμής το άρθρο 14.1 επιτρέπει μια τέτοια κατεξουσιοδότηση να υιοθετηθεί χωρίς την έγκριση του ε, Κοινωνικού Ταμείου. Ο κανονισμός που υιοθετήθηκε λοιπόν πέρσι δεν αλλάζει αυτή τη στιγμή το βασικό κομμάτι του κανονισμού έχουμε το εύρος του ορισμού ε, των ε, τυποποιημένων κλιμάκων μονοδιαίου κόστος ε, και των καταποκοπή ποσών τα οποία υιοθετήθηκαν πέρσι. Μονάχα τα παραρτήματα έχουν προσαρμοστεί διότι η Κομισιόν συνεχίζει να συνεργάζεται με, τα, με τις υπηρεσίες των κρατών μελών για να μπορέσει να αναπτύξει αυτές τις απλοποιημένες, τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστος και θα συμφωνήσουν σε προσαρμογές αργότερα. Ο κανονισμός πέρσι αναφερόταν στη Σουηδία και στη Γαλλία, ενώ αυτή τη στιγμή προσθέτουν, προτείνουμε ένα παράρτημα το οποίο περιλαμβάνει το Βέλγιο, ...και καθώς επίσης και ένα πρόγραμμα για την Τσεχία. Όπως ε, προανέφερα, δεν υπάρχει καμία αλλαγή όσον αφορά τα άρθρα Έχουμε εργαστεί στενά με το Βέλγιο και την Τσεχία για να επιτευχθεί αυτό το παράρτημα και αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με την Ιταλία, τη Μάλτα, τη Γερμανία, τη Σλοβακία και τις κάτω χώρες για περαιτέρω τροποποιήσεις ε, του κανονισμού με μέσα στη φετινή χρονιά, οπότε ίσως να συναντηθούμε και πάλι το φθινόπωρο με μια άλλη τροποποίηση του κανονισμού, όπου θα προσθέσουμε κάποια ακόμα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρουσίαση σχετικά με το περιεχόμενο του παραρτήματος. Αρχικά όσον αφορά την ε, Τσεχία έχουμε ε, πέντε ε, μοναδιαία κόστη, τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις δράσεις που έχουν ως στόχο τους την αύξηση της υποστήριξης ε, για τις υπηρεσίες υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, νηπιαγωγείων. Το πρώτο αφορά την υποστήριξη της απασχολησιμότητας ε, και στόχος ε, της κάλυψης αυτής της δράσης σχετίζεται με τη δημιουργία χώρων ε, σε υπάρχουσες αλλά και νέες εγκαταστάσεις νηπιαγωγείων, την βελτίωση των εγκαταστάσεων και το ποσό είναι στα 160 εκατομμύρια ε, τσεχικές κορώνες. Τα κόστη καλύπτουν τους υπολογισμούς ε, για το μοναδιαίο κόστος με βάση τις στατιστικές, ε, τις έρευνες της αγοράς ε, και μερικές φορές η όλη διαδικασία παίρνει κάτι παραπάνω. Δεν θα μπω όμως σε λεπτομέρειες. Βλέπετε τα πέντε ε, πλαίσια 1,6 εκατομμύρια κορώνες θα καλυφθούν σε αυτό η, η αλλαγή υπαρχουσών δομών 1,6 εκατομμύρια η ε, κάλυψη ε, νηπιαγωγείων εκεί θα υπάρχει μια υποστήριξη για 6 μήνες ανά και θα, έρθει και πάλι, θα ανέλθει και πάλι στα 1,6 εκατομμύρια Επίσης ένα άλλο ε, πρόγραμμα σχετικά με την καλή παροχή υπηρεσιών προ τα παιδιά, 1,8 εκατομμύρια. Δεν είναι, είναι λάθος ε, στην παρουσίαση αυτό, δεν είναι σε ευρώ, αλλά είναι σε κορώνες το ποσό. Για το Βέλγιο τώρα, το πλαίσιο δράσης αφορά δύο, ε, δύο σημεία που αφορά την εκπαίδευση που θα οδηγήσει στην απασχόληση καθώς επίσης και την επαγγελματική κατάρτιση που οδηγεί σε εξέβριση εργασίας αλλά με πιο γενικότερο τρόπο. Τα κόστη βασίζονται σε ε, αποδείξεις που έχουμε ήδη ε, με βάση την ε, Φλαμανδία διότι αυτό θα αναφερθεί μονάχα στο σχέδιο δράσης για τη Φλαμανδία τα ποσά θα πληρωθούν μονάχα όταν έχουμε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα, οπότε το άτομο ε, το οποίο θα λάβει τη συγκεκριμένη ε, κατάρτιση θα πρέπει να τα καταφέρει και το Βέλγιο δεν βλέπει κάποια προσαρμογή πάνω στα ποσά τα οποία έχουν συμφωνηθεί. Το η μεμονωμένη εκπαίδευση της επιχείρησης που σημαίνει ότι ε, κάποιο άτομο από το, ε, δημόσιο, ε, το δημόσιο θα λάβει εκπαίδευση και αυτό θα ολοκληρωθεί με ένα συμβόλαιο για το συγκεκριμένο άτομο στη συγκεκριμένη εταιρεία και προβλέπονται ε, περίπου, ε, 9.000 περίπου ευρώ Ενώ όταν υπάρχει εκπαίδευση που προβλέπεται από τις δημόσιες υπηρεσίες, η διαδικασία είναι μεγαλύτερη. Αρχικά θα πρέπει να υπάρχει ταυτοποίηση των συγκεκριμένων ανθρώπων, ε, θα πρέπει να, βρούμε το, να καταρτήσουμε το προφίλ τους, ποιες είναι οι ανάγκες τους, ε, τι οι δεξιότητες μπορούν να λάβουν, τι εκπαίδευση χρειάζονται και στη συνέχεια θα τους βοηθήσουμε ώστε να βρουν εργασία. Το ποσό λοιπόν για ένα άτομο προβλέπεται στα 8.466 ευρώ κατά το φλαμαδικό πρόγραμμα προβλέπει να ξοδεύσει 100 εκατομμύρια του συνολικού τους ε, προϋπολογισμού σε αυτό. Αν έχετε λοιπόν ερωτήματα είμαι διαθέσιμη. Thank you for... για την ενημέρωση. Η κυρία Σαρτιέ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή και την αγαπητή Αντριάννα που με τόση σαφήνεια παρουσίασε αυτό το θέμα, την τροποποίηση του κατεξουδότησης κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Προσυπογράφω πλήρω τα όσα μας παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς πρόκειται για απλούστευση και ταυτόχρονα για ενίσχυση των επιτευγμάτων χωρίς να αλλάξει η ουσία του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο στόχο έχει την αποτελεσματικότητα του ή άλλους. Άρα όποιο προσπάθει προς την αποτελεσματικότητα θα την υποστηρίξουμε και σας ευχαριστούμε για τις τροποποιήσεις αυτές που στηρίζουν τη δική μας βούληση να υποστηρίξουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, να το υπερασπιστούμε, να, το, να παρατηρούμε τη διάρκεια ζωής του. Δύο λόγια μόνο για να είναι απόλυτα σαφή η κατάσταση για τους πάντες. Πολύ καλά να παρουσιάζονται οι τροποποίησεις των αφορούν ε, συγκεκριμένα πρόγραμμα της Τσεχίας σε κορώνες τσεχικές, αλλά για μας καλό θα ήταν να βλέπουμε και ένα ισοδύναμο σε ευρώ. Γιατί δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι σημαίνει σε οικονομικούς όρους. Θα μας διευκόλυνε πολύ λοιπόν στην ανάγνωση των προτάσεων, αν είχε η Επιτροπή αυτή τη δυνατότητα. Και την ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ εσείς. Θα συμφωνήσω με την κυρία Μωρέν Σαρτιέ Καλό θέλω να έχουμε τα ποσά σε ευρώ. Αυτές οι 56 κορώνες παιδί είναι 2 ευρώ από ό,τι βλέπω, από ό,τι ξέρω εγώ. Αν μας δίνατε λοιπόν τα στοιχεία σε ευρώ, τουλάχιστον θα μπορούσαμε να κάνουμε μια αντιστοίχηση. Την έχετε ετοιμάσει την παρουσίαση αυτή διαθέσιμη, μπορείτε να μας την διαθέσετε. Είναι πολλές πληροφορίες, πολύ χρήσιμες. Θα χρειαστεί λίγο πιστός χρόνος για να τις εμπεδώσουμε. Θα ήθελα τη δυνατότητα λοιπόν να διαβάσω τη μελέτη. Καλώ ευχαριστώ. Η Επιτροπή μπορεί να δώσει τις ε, πληροφορίες σε ευρώ καταρχάς και τα άλλα στοιχεία που σας ρώτησαν. Δεν έχω ακριβή ε, ισοτιμία. 56 κορώνες είναι όντως περίπου 2 ευρώ αλλά αυτό είναι μια λύση που έχει εξευρεθεί μέσα με το κράτος μέλος. Σε κατεξοδότηση πράξη πάντα μπορούμε να στέλνουμε την επικαιροποίηση σε μονάδες σε κόστος ευρώ. Αλλά είναι αναγκαστικό αυτή η κατεξοδότηση πράξη να εγγράφεται σε, ισοτι... σε νόμισμα εθνικό. Γιατί έτσι γίνεται η χρηματοδότηση από το κοινωνικό ταμείο. Τα σημειώνω πάντως. Θα σας ενημερώσουμε με τον κατάλογο των ε, ε, του κόστους αναμονάδα και σε ευρώ και στο προσεχές παράρτημα εάν πρόκειται για κράτος που δεν έχει χρήση του ευρώ θα σας παρουσιάσω και σε ευρώ τους υπολογισμούς και όντως το είναι η απλοποίηση δηλαδή να μην χάνουμε πολύ χρόνο στους ελέγχους στην εξέβρεση λαθών παρατυπιών λογιστικού χαρακτήρα και να μπορούν οι αρχές διαχείρισης να βλέπουν ότι έχει επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα πριν κάνουν τις πληρωμές. Αυτός είναι ο στόχος της απλοποίησης και γι' αυτό έχουμε τις εντατικές συνομιλίες με τα πέντε κρατημέλη και περιμένουμε να συμμετάσχουν και άλλα αργότερα. Καλώς, ευχαριστώ. Μας αρέσει πολύ και μας η απλοποίηση. Σε ευρώ πάντως θα ήταν καλύτερο για να καταλάβουμε γιατί κλίμακα μιλάμε εμείς ως πολιτικοί. Σας ευχαριστώ, χρήσιμες πληροφορίες. Ιδιαίτερα υποστηρίζουμε το Ταμείο και την καλύτερη δυνατή χρήση του. Προθεσμία για την ε, Επιτροπή Απασχόλησης, για την ε, ε, κατάθεση αντιρρήσεων είναι 22 Απριλίου στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έκφραση αντιρρήσεων έως τις 18 Μαΐου. Πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ταμείο ε, Παγκοσμιοποίησης. Και η κυρία Χάρκιν έχει το λόγο. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Um, Η έκθεση αυτή για την προστιθέμενη αξία του Ταμείου για την παγκοσμιοποίηση λαμβάνει υπόψη την αρχική μορφή του κανονισμού, τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν πρόσφατη το 2014. Εξέτασα πολλά έγγραφα ε, για την έκθεσή μου, την έκθεση του, ε, ελεγκτικού συνεδρίου και θα παρατηρήσατε επίσης ότι σήμερα η Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κυκλοφόρησε μια νέα έκθεση. Ε, εγώ χρησιμοποίησα λοιπόν κάποιες προτάσεις, είναι μια εξαιρετική έκθεση νομίζω ότι συμπληρώνει τις ε, προτάσεις ε, αξιολόγησης εξ εκ των υστέρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω στα πλαίσια της πρότασής μου είναι να αξιολογήσω τις αλλαγές που, άλλα, που έγιναν στον τομέα της παρέμβασης από το 1500, τον διαφορετικό χρονισμό από 24 αρχικά μήνες σε 5 μήνες, τα θέματα της συγχρηματοδότησης από 50 σε 65, μετά σε 50 και τώρα σε 60, από 500 εκατομμύρια θα έλεγα κατέτος 150 και φυσικά και το θέμα Όταν γίνεται σαν παράδειγμα μια μορφή απολύσεων στις χώρες, αυτή τη στιγμή οι χώρες καταθέσουν αίτηση με, με ποια ταχύτητα ανταποκρίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουν σημασία βέβαια αυτές οι λεπτομέρειες τόσο πολύ όσο τα δικά σας σχόλια πάνω σε αυτά. Υπάρχουν ορισμένες ιδέες οι οποίες νομίζω είναι σημαντικές ένα από τα σημεία τα οποία εγώ υποστηρίζω και είναι κάτι το σχετικά καινούριο είναι ότι δεν θα πρέπει το Ταμείο αυτό να αντιμετωπιστεί σαν ένα μέσο αντιστάθμισης των εμπορικών και οικονομικών στρατηγικών. Σε κάποια φάση η Επίτροπος Μάλστρομ είπε ότι αυτά είναι θέματα εμπορικών συμφωνιών και μας είπε ότι όταν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στον τομέα της απώλειας θέσεων απασχόλησης, ε, πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιας και ο προϋπολογισμός μειώθηκε κατά τα 2 τρίτα και μιας και υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα σε πάρα πολλές περιοχές, ε, προφανώς η παρέμβαση της Επιτροπής δεν μπορεί ουσιαστικά να αλλάξει. Η πρόταση της Επιτροπής είναι, θα έλεγα, καλή. Δείχνει τον τρόπο με τον οποίο έχει χρησιμοποιήσει τα ποσοστά της ε, πάνω από 100%. Έχει εξαντλήσει και υπερβεί τα όρια. Και υπάρχουν λόγοι για αυτό το πράγμα Nonetheless, I think we do need accurate figures. So uh, the point is that if the, if the uh, όταν ένα κράτος μέλος ζητάει την παρέμβαση, ζητάει ας πούμε μια παρέμβαση για 500 εργαζομένους. Μετά βέβαια μπορεί να αλλάξει το, ποσοστό, το ποσό αυτό και να γίνουν και άλλες εταιρείες να θυγούν και να είναι 520. Αυτό σημαίνει επανυπολογισμό ουσιαστικά και υπέρβαση του 100% ενώ αυτό δεν ισχύει και παραμένουμε στα αρχικά επίπεδα. Ε, τώρα για την επαναπασχόληση των εργαζομένων προφανώς ε, σε σχέση με την παρέμβαση του Ταμείου δεν είναι κάτι το σημαντικό. Όμως ψυχολογικά βοηθά το Ταμείο αυτό. Έχοντας μιλήσει με αυτούς που ωφελήθηκαν από το Ταμείο αυτό Νομίζω ότι αυτό που μου είπαν ήταν το παρηγορητικό του, θα έλεγα, στοιχείο. Ε, τα ποσοστά εφαρμογής ε, είναι ένα θέμα από 3 μέχρι 110% με μέσο όρο 55%. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να επανεξεταστεί. Είναι ένα θέμα που έθεσε και το ελεγκτικό συνέδριο. Νομίζω πως ένα από τα πράγματα το οποίο έχει ουσιαστικά αλλάξει από τη δημοσίευση της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου είναι ότι τώρα τα κράτη-μέλη ε, προσφεύγουν στο ταμείο αυτό άμεσα μετά από την αίτηση προς την Επιτροπή. Ενώ παλιότερα μέχρι τώρα δεν το έκαναν αυτό και οι εργαζόμενοι έμεναν σε εκκρεμότητα 3-6 μήνες ή και περισσότερο πριν μπορέσουν να ενταχθούν στο ταμείο αυτό. Οι αρχικοί αριθμοί λοιπόν είναι, δεν φτάνουν στο 100% γιατί πολλοί από τους εργαζομένους ε, είχαν ενταχθεί σε άλλα συστήματα. Τα κράτη-μέλη επίσης δεν θα πρέπει να θέτουν ποσοτικούς στόχους επανένταξης σε αυτή τη φάση. Δεν είναι λάθος αυτό. Διαβάζοντας τις λεπτομέρειες της έκθεσης, βλέπω ότι τα δεδομένα τα οποία παίρνουμε δεν είναι τα κατάλληλα έτσι ώστε να αξιολογήσουμε σωστά την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία που παίρνουμε από τα κράτη-μέλη και χωρίς να επιβαρύνουμε γραφειοκρατικά τις απαιτήσει, πρέπει να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε καλύτερα ε, ε, το ποσοστό ε, επανένταξης. Και το ελεγκτικό συνέδριο απαιτεί από τα κράτη-μέλη να δουν τι δεδομένα θα χρησιμοποιήσουν για να δείξουν τα μέτρα τα οποία θα θέσουν σε εφαρμογή. Κατάρτιση και όχι αναζήτηση θέσης απασχόλησης. Εμφύσιση επιχειρηματικότητας ή το λεγόμενο mentoring καθοδήγηση δηλαδή. Λοιπόν, είναι πολλά τα στοιχεία που ζητάμε από τα κράτη-μέλη, πρέπει να τα εξετάσουμε προσεκτικά και να δούμε ακριβώς πώς ε, θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Να πούμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διαφοροποιήσουν ανάμεσα στις παρεμβάσεις του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης και του ε, Κοινωνικού Ταμείου. Απαιτούνται επίσης τακτικές εκθέσεις αξιολογήσεις εμπειρογνωμόνων και θα πρέπει να δούμε ακριβώς ε, πώς συγκρίνεται το νέο αυτό ταμείο με τις προηγούμενες δράσεις του και παρεμβάσεις του. Νομίζω ότι μαθαίνει κανείς από τα λάθη και τις επιτυχίες του. Κάποια τελευταία σημεία τα οποία κυκλοφόρησαν από τότε που ήδη συνέγραψα την πρότασή μου μετά από συναντήσεις και τα λοιπά. Ξέρω ότι οι συνάδελφοι θα έχουν να πούν πράγματα, αλλά τελειώνω. Ξεκαθαρίστηκε σε μένα ότι υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στον βασικό ρόλο του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης, για τους απολυμμένους δηλαδή, και την κάλυψη των αναγκών ευρύτερα. Οι ανάγκες ε, είναι στα πλαίσια μιας διαφορετικής προοπτικής και πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη και στα πλαίσια της λειτουργίας του ταμείου αυτού και στα πλαίσια της αξιολόγησης της λειτουργίας και θα συμφωνήσω με αυτό. Είχα επίσης ανταπόκριση καλή από τον κόσμο με τον οποίο μίλησα ότι θα πρέπει να παραμείνει τον στο εσωτερικό του ταμείου αυτού. Θα πρέπει να δούμε ποιοι άλλοι εταίροι μπορεί να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο προσπαθώντας έτσι ε, ώστε οι νέοι να καλύπτονται από το Ταμείο αυτό ε, και να καλύπτονται και από άλλους εταίρους που είναι ήδη δραστήριοι στον τομέα αυτό, ομάδες πρωτοβουλίας τοπικές κτλ. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να συνδυάζουμε ε, διαφορετικά μέτρα όπως το Νίτσα με το ταμείο αυτό. Ένα από τα θέματα τα οποία τέθηκαν τον προηγούμενη φορά που συζητήθηκε είναι το 25% για τις επιλέξιμες δράσεις. Κινητικότητα, επανακατάρτιση και ε, τοποθέτηση σε νέες θέσεις. Νομίζω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι με τους οποίους ε, ε, ε, συζήτησα μου ζήτησαν να μην αλλάξουμε το θέμα των ποσοστών. Τελειώνω λέει για τρίτη φορά η ομιλήτρια. Το άρθρο 4 είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό άρθρο. Είναι η εξαίρεση από τα κριτήρια εφαρμογής. Πήρα πολλά σχόλια και συζήτησα το θέμα αυτό με πολλούς άλλους συναδέλφους Πολλοί μίλησαν για μείωση των αριθμών, των ποσοστών και την πρόταση αυτή την είχαμε δεχτεί. Αυτό όμως το οποίο έχει σημασία είναι να προσπαθήσουμε να δούμε αν είναι κάτι το συμβατό με τον κανονισμό. Εγώ είδα το θέμα των αιτήσεων μέσω ε, για το ταμείο αυτό ε, από τότε που άλλαξε ο κανονισμός. 25 ήταν οι αιτήσει ε, και ε, ένα μεγάλο ποσοστό αφορά το άρθρο 4β για επιχειρήσεις κάτω των 500 εργαζομένων. Για το Βέλιο ε, υπήρξε μια περίπτωση 5.511 εργαζομένων. Μια άλλη αίτηση 939, 401 και 257. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ευελιξία η οποία υπάρχει στο εσωτερικό του κανονισμού για να καλύψουν θα έλεγα τις διαφορετικές μορφές απολύσεων μαζικών απολύσεων. Ένα από τα θέματα που πρέπει να τεθεί εδώ είναι ότι οι μικρομεσαίες και οι εργαζόμενοι στις μικρομεσαίες δεν καλύπτονται καταλήλως από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Ως εκ τούτου λοιπόν έκανα την πρόταση και ελπίζω να με στηρίξετε εδώ ότι όταν τα κράτη-μέλη καταθέτουν μία αίτηση ε, για μία σειρά επιχειρήσεων και για ένα συγκεκριμένο τομέα, οι κανόνες είναι σαφείς εδώ, ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προσφέρει έναν κάποιο πίνακα με επιμέρους ε, δυνατότητες για να καλυφθεί ο υψηλός αριθμός. Γιατί αλλιώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σε μια ακόμη φορά μειονεκτική θέση. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα κριτήρια ε, παρέμβασης, να δούμε πώς θα λειτουργήσει σωστά το 4β και τέλος, ε, όπως έχω πει τρεις φορές μέχρι τώρα, ε, θα ήθελα να πω ότι Εμείς θα τα δούμε όλα αυτά με πάρα πολύ προσοχή έτσι ώστε να μην υπάρξει ιδιαίτερη γραφειοκρατική επιβάρυνση και άγχος. Πήρα ένα email από μια επιχείρηση κρατική η οποία καλύπτεται από την κρατική ομπρέλα εν πάση περιπτώσει αυτό που στην Ιρλανδία ονομάζουμε ημικρατική που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση και μας είπαν ότι υπάρχουν, ε, μπορεί να έχει κανείς τέσσερις ομάδες ελεγκτών που να ελέγχουν τα ίδια στοιχεία και να καταλήγουν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Απαιτείται λοιπόν τα διάφορα επίπεδα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των διαδικασιών αυτών να έχει την δυνατότητα επανελέγχου και επαλήθευσης των στοιχείων που να καλύπτουν το σύνολο της διαδικασίας και όχι μία εταιρεία ορκωτών να καλύπτει ένα κλάδο και μία άλλη εταιρεία, ένα άλλο τομέα, μάλλον ένα άλλο τμήμα μιας κάποιας αίτηση. Νομίζω ότι αυτό περιπλέκει τα πράγματα. Δεν θα συνεχίσω άλλο και θα σας ακούσω αν έχετε κάτι να πείτε. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον κύριο Τσαμπασόγκος. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, παρακαλώ. Δεν θα είναι εύκολο να μιλήσω εγώ με την κυρία Χάρκιν, Πρόεδρε. Θα κάνω την μπορώ όμως. Ο κανονισμός αυτός δίνει απαντήνηση σε πολλά από τα ελλείμματα της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου, δίνει νέες προτάσεις, εισάγει νέες διατάξεις και θα πρέπει να δούμε και αν τα κράτη-μέλη είναι σε θέση να αξιοποιήσουν και την εμπειρία που έχουν αντλήσει από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, προκειμένου να ενισχύσουν την υλοποίηση, την εκτέλεση του προπολογισμού και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Το σχέδιο εκθέσεις προσφέρει μια πολύ καλή επισκόπηση των ζητημάτων ε, και των προβλημάτων βεβαίως χρηματοδότησης του παρελθόν και δίνει λύσεις για την καλύτερη αξιοποίηση του Ταμείου. Συμφωνώ ιδιαίτερως με την έκκληση πως θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη πρόβλεψη και ε, ως προς τις πολιτικές ε, επιλογές για την αγορά εργασίας, ώστε να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει από θε, εκ των υστέρων το πρόγραμμα προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα από την απουσία, από την κατάργηση θέσεων εργασία εκεί που έχουν παρεμβεί πολιτικέ επιλογέ. Επίση, υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, έχει μεγάλη σημασία. Το άρθρο 8 Δέλτα, παραδείγματι, για, την, ε, για τον εντοπισμό των ε, παραγωγών στην βάση της πυραμίδας, συμμετοχή διαφορών παραγόντων της οικονομίας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή συγκέντρωση αιτήματων από τον κατασκευαστικό και οικοδομικό και κυρίως την αυτοκινητοβιομηχανία και την αεροπνευπηγική και κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις. Με βάση λοιπόν τις θετικέ τάσεις που έχει εντοπίσει ε, για την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το τέλος των μέτρων και θα πρέπει να κοιτάξουμε την ενίσχυση των μέτρων αυτών και για το μέλλον. Ευχαριστώ. Thank you, shadow for the group. Μια και είμαι σκιώδης για τους θα σας πω και εγώ δύο λόγια. Αλλά ήταν πολύ καλή η έκθεση κυρίας Χάρκιν και έτσι έχω δυσκολία να βρω πολλά θέματα να αναπτύξω. Είναι καλή βάση λοιπόν για περαιτέρω συζητήσεις. Συζητήσεις που έγιναν στις συνεδριάσεις για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Τα θέματα που έχουμε συνήθως να συζητήσουμε με βάση την ημερήσια διάταξη έχουν να κάνουν με αναποτελεσματικές εμπορικές πολιτικές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Πρέπει να βρούμε συστήματα και συμφωνίε. χωρίς αυτόν. Δηλαδή να μην σημαίνει αυτό ότι δίνουμε με το ένα χέρι αυτό που έχουμε πάρει με το άλλο. Και μάλιστα με επιβάρηση γραφειοκρατική. Θα πρέπει να κάνει καλύτερε εξολογήσεις συνεπειών των εμπορικών τη συμφωνιών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να κάνει τις σωστέ επιλογές. Πρόκειται για, ένα, για μια κρίσιμη αφετηρία που θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλιστεί. Και ίσως χρειάζεται και να αναφέρουμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για την πρόβλεψη αλλαγών και αναδιαρθρώσεων που θα συστήσουμε εφέτος μεταξύ άλλων. Και μια και όλο και περισσότερα τα αιτήματα για το EGF δεν είναι αρκετό το πλαίσιο για να αντιμετωπίσει τις ε, συνέπειες των αναδιαρθρώσεων. Ίσως η κυρία Χάρκιν έχει κάποιες προτάσεις καλύτερες να μας κάνει, πάντως μπορούμε να συζητήσουμε πολλές διαφορετικές λύσεις. και ίσως μπορούμε να ζητήσουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις αναδιαρθρώσεις. Και μπορούμε να αξιολογήσουμε και να συστήσουμε τουλάχιστον την προοπτική. Η συνέπειση επίση, ο αντίκτυπο μάλλον του Ταμείου Παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να αξιολογηθεί καλύτερα. Ω προ την ε, διεύρυνση του πεδίου του Ταμείου Παγκοσμιοποίηση, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για τι συνέπειε, για τον αντίκτυπο και αν χρειάζεται εξωτερική αξιολόγηση. Όπως είπα, το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να αρχίσουμε να δίνουμε με το ένα χέρι αυτό που έχουμε πάρει με το άλλο και οι συστήσεις μας από τις συνεδριάσεις για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης αφορούσαν τις δυνατότητες να λαμβάνονται υπόψη και τα στοιχεία του εμπορίου. Και επίσης την αξιοποίηση του Ταμείου από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την αποτροπή καταχρήσεων ή καταστρατηγήσεων καλύτερα του Ταμείου από τις πολυεθνικές. Χρήσιμη, φαντάζομαι, ίσως και προκλητική η ερώτηση και ίσως θα ήταν καλό να την ε, λάβουμε υπόψη για τα περαιτέρω. Και ευχαριστώ δίνοντας το λόγο στην κυρία Μάκιντσάιρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω εκ μέρους ε, του σκιώδους του ECR που βρίσκεται ε, εκτός χώρας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 Ζητώ συγγνώμη που δεν βρίσκεται σήμερα εδώ. Αρχικά όμως ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χάρκιν για τη δουλειά της πάνω στην αναφορά που θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή και ισορροπημένη αναφορά. Χαιρετίζουμε λοιπόν από την πλευρά του ECR τη δυνατότητα ότι έχουμε αυτή την αναφορά διότι θεωρούμε ότι είναι σημαντικό όλες, ε, όλα τα έξοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ αυτού και του Ταμείου Παντοκοσμιοποίησης να εξετάζεται λεπτομερώς όσον αφορά την αξία των χρημάτων όπως ίσως γνωρίζετε, το ECR έχει κάποιες ανησυχίες όσον αφορά την προστιθέμενη αξία του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω κάποια γενικά σχόλια δεν θέλουμε να δούμε το Ταμείο να χρησιμοποιείται ως ένα μέσο το οποίο ε, χρηματοδοτεί τις εθνικές προσεγγίσεις και ούτε και υποστηρίζουμε ώστε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο το οποίο θα επεμβαίνει οπότε τα κράτη-μέλη έχουν αποτύχει να δράσουν. Και αυτό τονίζεται στην παράγραφο 18. Αρκετές εφαρμογές λοιπόν του, Ταμείου μπορεί να ε, αιτιολογηθούν ως, δικαιολογημένε, ως ε, δικαιολογημένες. Υπάρχουν πρόσφατες περιπτώσεις που μας ανησυχούν. Για παράδειγμα, η περίπτωση της Air France όπου η εφαρμογή μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ε, μια επιχορήγηση που δημιουργεί προβλήματα στην αγορά κάτι το οποίο αναφέρεται στα σημεία C και E. Όσον αφορά την επέκταση του κανονισμού, έχουμε κάποιες ανησυχίες ότι σε περίπτωση που το κάνουμε αυτό για να περιλαμβάνουμε τους αυτοαποσχολούμενους, τότε ίσως ε, να δίνουμε περιορισμένα ε, ποσά ε, πάρα πολύ αραιά, διότι έτσι θα περιορίσουμε την αποτελεσματικότητα του Ταμείου. Όμως, θα θέλουμε να πούμε ότι το ECR δεν υποστηρίζει την αύξηση του προϋπολογισμού του. Θα χαιρετίσουμε όμως τη δυνατότητα να εξετάσουμε μέσα με τα οποία το Ταμείο θα μπορεί να είναι πιο στοχευμένο και επικεντρωμένο για να μπορέσουμε να εξοδεύουμε λιγότερα χρήματα πιο αποτελεσματικά. Ο λόγος ε, για να διευρύνθει ε, ο σκοπός ε, του Ταμείου ε, όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες μας ανησυχεί. Το 2013 το ελεγκτικό συνέδριο έκανε ορισμένες παρατηρήσεις λύσεις οι οποίες αναφέρθηκαν στο νέο κανονισμό, όμως υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία υπάρχουν ακόμα. Για παράδειγμα, πάρα πολλά από τα μέτρα του Ταμείου θα μπορούσαν ε, να ε, αντιμετωπιστούν και μέσω του Κοινωνικού Ταμείου. Πολλά όμως, ε, κρατικά, πολλά όμως κρατημέλη επέλεξαν να το χρησιμοποιήσουμε και, θα, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να ενσωματώσουμε τους ε, στόχους ε, του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης στο Κοινοτικό Ταμείο και αυτό αναφέρεται στην αναφορά μου. Το ελεγκτικό συνεδρίο ανάφερε ότι τα υπάρχοντα δεδομένα δεν ήταν επαρκή για να μπορέσουμε να, για να αξιολογήσουμε τα μέτρα επανενσωμάτωσης των εργαζομένων και αυτό οφείλεται στην έλλειψη ε, δεδομένων για το συγκεκριμένο ζήτημα. Όταν δημοσιεύθηκε η συγκεκριμένη αναφορά το 2013 υπήρχαν ήδη διαπραγματεύσεις για ένα νέο κανονισμό του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης για την περίοδο 14-2020 και θα πρέπει να δούμε αν οι νομοθέτε μπορούν να οργαστούν πιο ε, αναλυτικά με το ελεγκτικό συνέδριο για το αν μπορούμε να προσθέσουμε ε, περισσότερα δεδομένα. Ενώ τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια για το έργο τη και ε, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε επικοδομητικά τις επερχόμενε εβδομάδες πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Link Boylan. Ευχαριστώ, δεν έχω μπροστά μου το όνομά μου. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, δουλειά της ε, και να επαναλάβω ε, τα σχόλια και θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις επιρροές της αποφάσεις στην αγορά εργασία θα ήθελα να προσθέσω ότι η Κομισιόν δεν θα πρέπει να προβλέπει μονάχα καλύτερα τις συνέπειες, αλλά θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της ε, εμπορικής της στρατηγικής η προστασία ε, των θέσεων εργασίας ε, στις διαπραγματεύσεις της. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να συμπεριλάβω είναι τα μαθήματα τα οποία διδαχθήκαμε από την εφαρμογή των δυνατοτήτων του Ταμείου στην Ιρλανδία, τη χώρα μου, ε, μία από τις σημαντικότερες ανησυχίες εκεί πέρα είναι το γεγονός ότι ε, πάρα πολλά ε, μεγάλα ποσά επιστρέφονται στην Κομισιόν στο Δουβλίνο μιλάμε για 4 εκατομμύρια, για περίπου για ένα ποσό 4 εκατομμυρίων τα οποία θα επιστραφούν σε περίπτωση που δεν θα πανηθούν και θα πρέπει να γίνει ένα αίτημα για, τις, για την ελευθερία πληροφόρησης. Πιστεύω λοιπόν ότι κάτι το οποίο μπορεί να συμπεριληφθεί είναι να υπάρξει μια αυξημένη διαφάνεια στη διαδικασία αλλά και υποστήριξη για τους ε, νέους και χαιρετίζω επίσης τα σχόλια της εισηγήτριας για την ανάγκη διαμυρισμού εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών τα κράτη λοιπόν τα οποία περιόρισαν ε, τα έξοδά τους ε, θα μπορούσαν να διδάξουν πολλά στην Ιρλανδία για παράδειγμα. Οι Κομισιόν ε, και οι υπεύθυνε υπηρεσίε θα πρέπει να ενημερώνονται και θα πρέπει να περιλαμβάνονται και αναφορές σχετικά με τις δαπάνες καθώς επίσης ε, και θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με το πώς να αποφεύγονται τα ε, υπερβολικά έξοδα. Σχετικά με τις ανάγκες είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τα μέτρα τα οποία ε, ελήφθηκαν και θα θέλουμε να δούμε μια ανεξάρτητη αξιολόγηση για το θέμα αυτό που θα εξετάζει ιδιαίτερο στην συμμετοχή του ΜΙΤΣ και θα ήθελα η συγγήτρια ε, να περιλάβει ε, και την κοινωνία ε, στο θέμα διότι εκτός από τις κρατικές υπηρεσίες υπάρχει ένα ολόκληρο σώμα θα λέγαμε ανθρώπων οι οποίοι είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν πάνω στη διαδικασία θα με ενδιέφερε να μάθω διότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην Ιρλανδία. Η συγκήτρια ανέφερε ότι υπάρχουν αρκετές χώρες οι οποίες ξεκινούν τη διαδικασία όταν έχουν αποστείλει την αίτηση χωρίς να περιμένουν την έγκριση. Δεν, ξέρω, νομίζω ότι κάτι τέτοιο ισχύει στην περίπτωση της Ιρλανδίας. Ένα άλλο θέμα το οποίο αναφέρθηκε είναι τα πολυετή προγράμματα κατάρτισης τα οποία θα πρέπει να παρέχονται μετά τη λήξη του ε, προγράμματος εφόσον η έναρξη του προγράμματος είναι μέσα στο χρονικό πλαίσιο του προγράμματος η διαδικασία και πάλι όμως ε, πάρα πολλά τέτοια ε, προγράμματα είναι τριετή και λαμβάνουν χρηματοδότηση μόλις για δύο χρόνια. Και πάλι ευχαριστώ την εισηγήτρια για το έργο της και θα χαρώ να συνεργαστώ μαζί της καθώς επίσης και με τους ευρωβουλευτές από όλες τις ε, ομάδες για να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η Μόνικα δεν είναι εδώ, η Τζιν είναι. Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ αντικαθιστώ τη Μόνικα που είναι απούσα. Μου έδωσε όμως τις σημειώσεις της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την Χάρκιν για μια πολύ πλήρη εισαγωγή που με βοήθησε ακόμα και μένα να καταλάβω το τι σας διαβάζω στην παρούσα φάση. Η Μόνικα λέγει ότι γενικά μπορούμε να υποστηρίξουμε πολλές από τις ιδέες της hacking. Ένα από τα θέματα ήταν το θέμα των αποζημιώσεων. Είναι ένας τομέας ο οποίος πρέπει να συζητηθεί ακόμα περισσότερο. θα πρέπει να μειωθεί το ανώτατο όριο του 35%. Εδώ είναι κάτι το οποίο νομίζω όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Συμφωνώ επίσης με αυτούς που λέγουν ότι πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα μέτρα τα οποία επιτρέπει να ληφθούν το Ταμείο αυτό να μην αποκλείουν αντίστοιχες παρεμβάσεις από πλευράς των υπηρεσιών των κρατών μελών και πρέπει να υπάρξει εδώ συμπληρωματικότητα. Πρέπει να τα διευκρινίσουμε αυτά, ιδιαίτερα στα πλαίσια του 7β, έτσι ώστε δράσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των επιχειρήσεων και των κρατών μελών να μην χρηματοδοτούνται από το Ταμείο. Θα επανέλθουμε σαν σκιώδης για το θέμα το οποίο τέθηκε για τις μικρομεσαίες. Υπάρχει έτσι και αλλιώς πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση και με την αλυσίδα της, ε, των προμηθειών κτλ. Ε, και είναι μια διάσταση η οποία πρέπει να καλυφθεί, ειδικά για τις μικρομεσαίες, επίσης ε, για τον λογιστικό έλεγχο. Οι λογιστικοί έλεγχοι οι οποίοι γίνονται πρέπει να είναι αποτελεσματικοί και να μας δίδουν τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται. Και η πολλαπλότητα των λογιστικών ελέγχων δεν βοηθά πάντα. Είναι κάτι το οποίο έχουμε υπόψη μας και σε άλλους τομείς. πρέπει να το εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος. Αυτά. Ατζία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την συνάδελφο Χάρκιν για την αρχική της πρόταση επί της οποίας έχουμε κάποιες παρατηρήσεις της διαιρώ δύο κατηγορίες, την τεχνική κατηγορία και την πολιτική. Η πρώτη, αυτό το οποίο φαίνεται σαφές εδώ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη δεν μας έχουν δώσει τους ποσοτικούς στόχους που να επιτρέψουν να θέσουμε ε, θα έλεγα ξεκάθαρα όρια για την επανένταξη των εργαζομένων και αυτό δημιουργεί σύγχυση. Έχει υπάρξει σαφώς σύγχυση ανάμεσα στην χρήση του συγκεκριμένου ταμείου, του κοινωνικού ταμείου και όλα αυτά δεν βοηθούν να ξεκαθαριστούν ε, θα έλεγα οι διαδικασίες. Έχει σημασία λοιπόν εδώ να προχωρήσουμε σε μια πρώτη ανάλυση. Δεύτερον, η Επιτροπή εκτιμά θετικά ότι το ότι το 50% τουλάχιστον επανένταξης είναι ένας θετικός στόχος. Χωρίς όμως να γίνεται εδώ η διάκριση σε ποιο βαθμό από τους εργαζομένους έχουν επωφεληθεί από το Ταμείο και πόσοι άλλοι έχουν επωφεληθεί αποκλειστικά από το Κοινωνικό Ταμείο. Και εδώ δημιουργείται σύγχυση ένα τρίτο σημείο είναι συνολικά ποιες είναι οι αιτήσει για την χρήση του ταμείου αυτού και ποιες είναι οι εκτιμήσεις επί της ουσίας οι οποίες γίνονται από την Επιτροπή. Πόσες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποκλείονται διότι δεν εντάσσονται στις προϋποθέσεις. Προέρχομαι από μια χώρα όπου οι αριθμοί πρόσβασης αναεργαζόμενο στο Ταμείο δεν είναι κάτι το δυνατό γιατί δεν φτάνουμε στο κατώτατο όριο, στα ελάχιστα όρια για τη χρήση του ταμείου αυτού. Στις περισσότερες περιπτώσεις προβλέπεται η χρήση του κοινωνικού ταμείου. Είναι κρίμα λοιπόν που αποκλείονται οι διαφορετικές δυνατότητες και αυτό το οποίο παραμένει για να λειτουργήσει υπέρ των ανέργων είναι ένα ελάχιστο οικονομικό ε, διαθέσιμο. Τώρα, για την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου του 2013, η διάρκεια έγκρισης μιας αίτησης είναι 41 εβδομάδες. Αυτό είναι κάτι το οποίο οδηγεί στις περισσότερες επιχειρήσεις να προσφεύγουν στο κοινωνικό ταμείο μέσω των περιφερειακών οργάνων του που ανταποκρίνεται ε, σε πιο, με πιο υψηλές ταχύτητες. Πρέπει να αναζητήσουμε λοιπόν λύσεις όχι μόνο πιο αποτελεσματικές. Ένας εργαζόμενος 50 ετών που χάνει τη θέση του δεν μπορεί εύκολα να βρούμε κάποιο μέσο όπως η εγγύηση για τους νέους ή η αυτόματη προσφυγή σε μια διαδικασία κατάρτισης. Είναι άνθρωποι με ικανότητες, με ε, ε, που είναι οικογενειάρχες ε, στο εσωτερικό μιας επιχείρησης, ε, δούλευαν επί μακρόν και πρέπει να υπάρξουν ad hoc για τους ανθρώπους αυτούς και συνοδευτικά μέτρα ενίσχυσης ε, που συνοδεύουν τη διαδικασία κατάρτισης γιατί κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του επανακατάρτισης πρέπει να έχει και χρήματα το 4 ευρώ την ώρα που παίρνουν κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας κατάρτισης προφανώς δεν μπορεί να το κάνει ένας οικογενειάρχης. Όλα αυτά λοιπόν είναι δεδομένα τα οποία μπορώ να σας τεκμηριώσω. Και όταν μιλάμε για ταμείο προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, αναφερόμαστε σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που κλείνουν λόγω της, του ανταγωνισμού των, εξ, των εκτός Ευρώπης επιχειρήσεων. Ένα άλλο ερώτημα τίθεται εδώ. Βλέπω ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις που είναι σε κρίση στην ουσία μετέφεραν την παραγωγή τους σε άλλες χώρες. Οι μετακινήσεις λοιπόν των επιχειρήσεων είναι κάτι που δεν λαμβάνουμε υπόψη. Απ' τη μία κρίνουμε το TTIP, από την άλλη την ε, παραχώρηση του καθεστώτος οικονομίας της αγοράς στην Κίνα. Μιλάμε για εκατομμύρια θέσεων εργασίας που θα χάσουμε. Πώς θα τις διαχειριστούμε με το Ταμείο Προσαρμογής. Πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε θέματα που θα θίξουν την Ευρώπη βραχυπρόθεσμα. Το Ταμείο αυτό λοιπόν δεν λαμβάνει υπόψη και τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες των νέων που είναι εκτός εργασίας και ένα τελευταίο στοιχείο βλέπω να υπάρχει μια κάποια αντίφαση. Από το 7 μέχρι σήμερα υπήρξε μια αύξηση των αιτήσεων προσφυγής στο Ταμείο. Από την άλλη έχουμε πάρα πολλές ε, παρατηρήσεις να κάνουμε στο ότι η επανατοποθέτηση αυτού ο οποίος έχει επανακαταρτιστεί και τα δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική για τους εργαζομένους διότι αυτό δημιουργεί πολλές φορές, συνοδεύεται από προβλήματα. Και όπως είπαμε οι μικρομεσαίες είναι εκτός, εμείς θα θέλαμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι, να καλύψουμε και τις μικρές επιχειρήσεις, πριν δηλαδή αναφερθούμε στο ταμείο αυτό και εξαντλήσουμε, πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις άλλες δυνατότητες ή μήπως η μοναδική εναλλακτική λύση που έχουμε είναι η συγκεκριμένη. οι επιχειρήσεις οι οποίες μετακινούν τις επιχειρήσεις τους αλλά έχουν πάρει κοινοτικά χρήματα πρέπει να τα επιστρέψουν τα χρήματα αυτά. Το να τσεπώνω τα κοινοτικά χρήματα της πιστώσης και σε ένα χρόνο να φεύγω αυτό είναι απαράδεκτο πρέπει να τα επιστρέψω διότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρώπη και εμείς σαν Επιτροπή Κοινοβουλευτική Απασχόλησης είμαστε κατά αυτών των απαράδεκτων πρακτικών. Θα στείλουμε τις ερωτήσεις αυτές γραπτά στη συνάδελφο για να τις λάβει υπόψη και θα συνεργαστούμε στα πλαίσια των συναντήσεων των σκιωδών. Ο κύριος Μαρτά. Ευχαριστώ. Ξέρουμε όλοι ότι αυτό το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση καθιδρύθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καταστροφικέ συνέπειε τη παγκοσμιοποίηση, καταστροφικέ για του εργαζομένου βεβαίω. Η ε, εξαφανιστή βέβαια θέση εργασία σπάνια, αντικαθιδαπονέ από νέε και η αγορά εργασία είναι πολύ δύσκολη για του ενέργου. Οι νέοι ιδιαίτερω αντιμετωπίζουν το φάσμα τη κινητικότητα, η δε πιο ηλικιωμένη το φάσμα της ανεργίας. Είναι γνωστό επίσης ότι πολλές περιοχές, ε, οι επιχειρήσεις που πλήττονται από την κοσμιοποίηση, είναι θύματα των εμπορικών πολιτικών, όπως είπε ο κ. που αποφασίζει το ευρωπαϊκό επίπεδο. Εσείς δηλαδή. Και αναφέρομαι στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, που έχουν ήδη συναυθεί, που βρίσκονται υπό διαπραγματεύσει μάλιστα με πολύ μυστικέ διαδικασίε και επίση των μελλοντικών με την Κίνα κτλ. που είναι κύριοι φόροι μαζικών απολειών θέσεων εργασία στην Ευρώπη. Με άλλα λόγια. Με άλλα λόγια. Πιστεύω ότι προσπαθούμε φιλότιμα να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες παγκοσμιοποίησης, αλλά όχι τις αιτίες της τις γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω. Και, και πρέπει να προσθέσω γνωστό ότι τα χρήματα αυτά φεύγουν από το Ταμείο Αποκοσμιοποίηση, αλλά όπω συμβαίνει τουλάχιστον στην Ελλάδα, δυστυχώ οι εργαζόμενοι δεν βλέπουν πότε τα χρήματα αυτά. Δεν ξέρω ακριβώ τι συμβαίνει. Υπάρχει ένα φαινόμενο εξάτμιση στο Ταμείο Προσαρμογή στην εντυπωσιακό. και συχνά υποστηρίζουμε εμεί ω Γάλλοι βουλευτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί ξέρετε ότι η Γαλλία είναι καθαρό χρηματοδότη κατά 8 δι ευρώ. Το να ψηφίζουμε λοιπόν αυτό το Ταμείο αποκοσμιοποίηση αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τη δυνατότητα να ανακτήσουμε τα χρήματα του Γάλλου φορολογουμένου. 22 δι διαθέτουμε, 12 μόλι ανακτούμε. Ευχαριστώ την κυρία Χάρκιν του των Λεχθέντων για τη δουλειά της. Ειλικρινή και, αντα... και Δεν κρύβεται πίσω από το δαχτυλό της κυρία Χάρκιν. Λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Και τελικά μας δει, λέει ότι δεν δουλεύει καλά το σύστημα. Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για την αξιολόγηση. Οι συνέπειες αντικτύπου είναι ασαφείς. Είναι πολλοί οι παρεμβαίνοντες και οι αξιολογήσεις, οι λογιστικές, οι λογιστικοί Τέσσερις για την Ιρλανδία, σε μια περίπτωση. Ποιος πληρώνει όλα αυτά τα γραφεία λογιστικού ελέγχου και ποιος λέει την αλήθεια. Ξέρετε πολύ καλά σε ποιον πάνε τα χρήματα. Τα είπε και η κυρία Στις μεγάλες πολυεθνικές που μετακινούνται προς άλλους ουρανούς και στους οποίους θα πρέπει να πούμε «Give me my money back». Δώστε μας πιο τα λεφτά. Αυτά έπρεπε να πούμε. Εκεί, πρέπει να πάνε τα χρήματα, ε, εκεί δεν πρέπει να πάνε τα χρήματα, αλλά στι μικρομεσαίες επιχειρήσει που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε τρεις αδέλφου ακόμη μετά την Επιτροπή και για το τέλος την κυρία Χάρκιν. Και επειδή δεν έχουμε τους διερμηνείς για πολλή ώρα ακόμα, θα σας παρακαλέσω να είστε σύντομοι, κυρία Ρενά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η αλήθεια δεν βρίσκεται ποτέ μέσα σε σχηματοποιημένη παρουσίαση των ριζοσπαστορακραίων. Ευχαριστώ την κυρία Χάρκιν για τη δουλειά της. Δεν έχω την ίδια ευρωπαϊκή εμπειρία με την κυρία Χάρκιν που παρακολουθεί εδώ και αρκετό καιρό την υπόθεση. Έχω εργαστεί από την άλλη πλευρά, δηλαδή την εγκατάσταση ε, κέντρων προσαρμογής, αναπροσαρμογής ε, στο Βέλγιο. Είπε η κυρία Χάρκιν ότι το Βέλγιο έχει αντιληφθεί καλά τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Φαντάζομαι ότι και εκείνη με κάποιο θετικό τρόπο βλέπει τον τρόπο λειτουργίας ως προς την αναπροσαρμογή του Βελγίου. Έναν τρόπο ο οποίο υλοποιήθηκε με την συνδρομή των κοινωνικών εταίρων, των δημοσίων υπηρεσιών και των ιδιωτικών εταίρων, συνδικάτων και και που επέτρεψε έτσι να καταλήξουμε σε μια διαρθρωμένη πρόταση για την αναπροσαρμογή, για την αναδιάρθρωση. Πάντως μπορέσαμε να θεσμοθετήσουμε μια σειρά από λειτουργίες και το γεγονός ότι ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες διέπονται από τον νόμο πλέον δεν επιτρέπει την παρέμβαση του αμείου. Άρα χρειάζεται να υπάρξει αυτή η λειτουργία της προσθετικότητας που ανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι το ότι, ήμασταν, ήμασταν στο κράτο ήταν ευαίσθητο σε θέματα κοινωνικά και ανάγκε των εργαζομένων. Μπορεί να σημαίνει ότι ζητούμε περισσότερα, αλλά έχουμε χαμηλότερα ποσοστά παρέμβαση, γιατί το μεγαλύτερο μέρο του κόστου καλύπτεται και από το ίδιο το κράτο και από τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Ίσως βέβαια, εάν όλοι έπαιρναν το ίδιο, να είχαμε καλύτερα αποτελέσματα να καλύπταμε περισσότερο τις ανάγκες των εργαζομένων σε τοπικό επίπεδο. Υπενθυμίζω και ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να κάνω μια διόρθωση για να βρεθεί σε μεγαλύτερη άνεση η Επιτροπή σχέση με τον κανονισμό, γιατί είχαμε συστήσει την για το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση στην αξιολόγηση, στην εσωτερική αξιολόγηση, μεσοπρόθεσμη ή, ή εξωτερική πάλι μεσοπρόθεσμη. Για να διευκολύνουμε λοιπόν την Επιτροπή, θα ήταν καλό να διευκρινιστεί αυτή η αξιολόγηση με το άρθρο 20 του κανονισμού. Μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση που αυτή τη στιγμή αφήνει ε, μια ασάφεια σε σχέση με την δυνατότητα για την Επιτροπή να προσφύγει σε εξωτερικούς ε, αξιολογητές. Εάν δεν αλλάξει το σχετικό άρθρο του κανονισμού, θα πρέπει η Επιτροπή να αιτιολογεί γιατί προσφεύγει σε εξωτερικό αξιολογητή. Ρόλος μας άλλωστε ως βουλευτών είναι να ε, παρακολουθούμε την ε, σωστή εφαρμογή των κανονισμών. Άρα είτε να το τροποποιήσουμε για να σας διευκολύνουμε ως προς τη ε, προσφυγή σε εξωτερική αξιολόγηση, είτε να παρακολουθούμε τις επιλογές σας. Για την πολιτική προσέγγιση τώρα το Ταμείο αυτή τη στιγμή έχει μόνο παρηγορητικό χαρακτήρα. Δηλαδή προσπαθεί να αντιμετωπίσει συνέπειες μόνο. Και δεν συμφωνώ με την Επίτροπο Μάλστρομ όταν στην νέα εμπορική στρατηγική New Trade Strategy, το έγραφα αυτό για τη νέα στρατηγική για το διεθνές εμπόριο, ε, λέει ότι γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν ε, πόλεις της συνεργασία και ότι αυτές ε, τις ε, Θέσει εργασία που θα χαθούν δεν έχει παρά να τις αποζημιώσει το Ταμείο για την παγκοσμιοποίηση. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε έτσι. Δεν μπορούμε να ξεκινούμε με τι εμπορικέ συναλλαγέ βλέποντα τα πάντα βέβαια μαύρο όπω έκανε μόλις τώρα ο κύριος Μαχτά. Αλλά θα πρέπει να αναλύουμε τι δυνατότητε του διεθνού εμπορίου σε θετικέ και σε αρνητικέ. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι μπορεί να υπάρξουν συνέπειε αρνητικέ σε κάποιου τομεί ή περιοχέ που μπορούν ενδεχομένως να έχουν και συνέπειες ως προς τις θέσεις εργασίας. Θα πρέπει μάλιστα να τις προλαμβάνουμε και να δίνουμε τα, μέτρα της αναπροσαρμογής, τα μέσα της αναπροσαρμογής για τις περιοχές και τους τομείς εκείνους που κινδυνεύουν περισσότερο από τους μηχανισμούς της παγκοσμιοποίησης. Αντίθετα λοιπόν από αυτό που προτείνει, που προβλέπει στην στρατηγική της για το Εμπόριο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει πιστεύω να διευρύνουμε τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση ώστε να προλαμβάνει μια σειρά από Έγινε λόγο για την αναγνώριση του καθεστώ οικονομία τη αγορά στην Κίνα. Υπάρχουν εκτιμήσει που αναφέρονται σε απόλυτα 250.000 θέσεων εργασία και αυτή είναι η καλή εκδοχή, μέχρι 3 εκατομμυρίων. Η πρώτη ήταν η εκτίμηση τη επιτροπή η δεύτερη των επαγγελματικών ενώσεων. Από 250.000 σε 3 εκατομμύρια θέσει εργασία μπορούν να χαθούν εάν αναγνωριστεί το καθεστώ οικονομία αγορά στην Κίνα. Ε, νομίζω πια ότι πρέπει και ο τομέα και οι περιφέρειες να εξασφαλίσουν μέσα για να προλάβουν κάποια δυσμενή εξέλιξη. Και δεν μιλούμε για 25.000 ευρώ που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Θα χρειαστούν περισσότερα μέσα ως πόροι, αλλά και ως δυνατότητες δράσης του Ταμείου για την παγκοσμιοποίηση. Επίσης, στην αξιολόγηση. Όταν γίνεται αξιολόγηση προς το ποσοστό επανυπολογισμού, όταν κλείνει μια επιχείρηση, ένα τομέα, ο επαναπροσδιορισμός μπορεί να οδηγηθεί σε πολύ, σημαντικές, σε πολύ σημαντικά ποσοστά ως προς την, το ποσοστό αναπροσαρμογής. Όταν έχουμε μία μονοτομιακή όμως περιοχή που κλείνουν όλες οι επιχειρήσεις λόγω της παγκοσμιοποίησης, το 80% επαναπροσδιορισμός είναι αδύνατο ποσοστό. Ούτε καν 50% δεν είναι δυνατόν, διότι το ολόκληρη περιοχή. Και εκεί νομίζω θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αυτή η πραγματικότητα περιφερειακού χαρακτήρα, δηλαδή μία μονοτομεακή περιφέρεια που ε, επλήγει λόγω της ε, μη βιωσιμότητας ενός τομέα. Και επίσης σήμερα το πρωί συναντήθηκα με εκπροσώπους του τοπικού εμπορίου που είναι και η προθήκη της Ευρώπης που έμεσα πλήττονται από απεριμώσεις ε, περιοχών και προωτούν γιατί ο τοπικός έμπορος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης λόγω των έμεσων συνεπειών της απερίμωσης μιας περιοχής. Πώς μπορώ να συνεχίσω να ζω σε μια περιοχή και να αναπτύσσω τοπικό εμπόριο όταν κάποιος τομέας έχει τελείως εξαφανιστεί από αυτήν. Αυτό λοιπόν πρέπει να το ενσωματώσουμε. Και όχι μόνο μικρομεσές ε, ή μεγάλες επιχειρήσεις σχετικές με ένα συγκεκριμένο τομέα, αλλά και τον έμπορο που μπορεί ε, επιχειρηματικά να βρίσκεται μακριά από το τομέα αυτόν θα μπορούσε να δώσει νέα ε, ζωή στην περιοχή. Και επίσης το 35% επί των εισοδημάτων, η παρέμβαση δηλαδή για τους ανέργους. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Κοσμιοποίηση βεβαίως δεν είναι εισοδηματικό εργαλείο για τον ε, άνεργο για εκείνον που έχει χάσει τη δουλειά του. Αλλά είναι πολύ πιο πρακτικό να δουλεύει κανεί με ανθρώπου και που έχουν χάσει τη δουλειά του, αλλά και που βρίσκονται σε συνθήκε φτώχεια. Δεν μπορούν, παραδείγματι, να προσφύγουν σε δανειοδότηση από τι τράπεζε. Εάν δεν μπορούμε να καλύψουμε λοιπόν το εισόδημά του, τότε ε, εμποδίζουμε και την τοπική ανάπτυξη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι χάνουν τα πάντα. Πρέπει να διατηρήσουμε λοιπόν μια ευελιξία ω προ τη δυνατότητα να λαμβάνεται υπόψη ένα ισοδηματικό κριτήριο για εκείνους που έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω, του Ευρωπαϊ... ε, λόγω της παγκοσμιοποίησης. Ευχαριστώ κυρία Μόνε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Χάρτινγκ για μια εξαιρετική δουλειά. Ε, γνωρίζει σε βάθος ε, το Ταμείο αυτό και γι' αυτό το λόγο οι γνώσεις που έχει για το θέμα από τη μία και η μεγάλη της ειλικρίνη από την άλλη καθιστά την πρότασή της ιδιαίτερο σεβαστή. Θα ήθελα για ένα θέμα να γνωρίσω την ουσία ενός θέματος το οποίο αγνοώ η ουσία λοιπόν για κάποια θέματα είναι άγνωστη. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί το ταμείο αυτό δεν την χάνει σωστής προώθησης. Έχω δει πάρα πολλούς υπουργούς στα κρατη να μην γνωρίζουν το ταμείο αυτό. Ενώ οι υπουργοί είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να διαφημίζουν αυτή την δυνατότητα σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμα και σε περιφερειακό επίπεδο επίσης ε, υπάρχει μια άγνοια ε, για ποιο λόγο, ίσως γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε την πρόθεσή του ή ίσως ε, θα πρέπει να επιλέξουμε μια διαφορετική λύση. Εγώ είμαι υπέρ του ταμείου αυτό, το παρακολουθώ από το 2007. Έχω δει ε, επίσης τις δυνατότητες που παρέχει στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους. Αν χρησιμοποιείται σωστά, Έχω ορισμένα παραδείγματα επικοδομητικά για την χρήση του ταμείου αυτού, ε, για τον εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων και για νέες γραμμές παραγωγής, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι που έχουν ανακατακαταχθεί έχουν ε, αποκτήσει μια νέα όφηση. Είμαστε ε, πέραν της φιλανθρωπίας, είμαστε πέραν του κοινωνικού ταμείου και ενώπιον μιας πραγματικής προστιθέμενης αξίας. Για τους ελέγχους, Μάριαν, ε, συμφωνώ. Θα πρέπει επίσης ε, να πούμε ότι το 6 αυτό της 100 είναι ιδιαίτερα χαμηλό το κόστος λειτουργίας δηλαδή αν δούμε πόσα επίπεδα ελέγχου υπάρχουν, γιατί θα έχουμε περισσότερους ελέγχους παρά ποσοστά κόστους λειτουργίας. Το τρίτο σημείο είναι τα ωφέλη τα οποία οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν από το ταμείο αυτό βλέπουμε ότι όταν εργαζόμαστε σε επίπεδο περιφερειακό ή όταν εργαζόμαστε σε επίπεδο τομέα συνολικά, ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολλές πολύ μικρές επιχειρήσεις που επωφελήθηκαν από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Η φαντουργία στην Πορτογαλία, ξυλία στην Ισπανία Εκεί μπορέσαμε οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες να ωφεληθούν. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνεχίζουμε να στηρίζουμε. Γιατί δεν πρέπει να είναι ένα ταμείο το οποίο να μην ωφελεί παρά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους εργαζομένους των μεγάλων επιχειρήσεων και οι εργαζόμενοι στις μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να τύχουν στήριξης για την ανακατάταξή τους στην επαγγελματική. Σύνεπως λοιπόν είμαι υπέρ του να βοηθήσουμε την εξέλιξη του ταμείου αυτού, να είναι αναγνώσιμη η εξέλιξή του και να ωφελεί τους εργαζομένους. Και γι' αυτό στηρίζω πλήρως αυτά τα οποία είπε η Μάριαν για την ανάγκη περισσότερης ευκρίνειας στον τομέα αυτό. Τέλος, μια ερώτηση θα ήθελα να θέσω σχετικά με το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης και την οικονομική κρίση. Θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε, Μάριαν, κάποια εμπόδια στην υψηλότατη στιγμή της, ε, της ε, χρηματοοικονομικής κρίσης. Νομίζω ότι σε ορισμένους τομείς σήμερα η έννοια της κρίσης πρέπει να είναι πάντα στο νου μας, γιατί αλλιώς θα συγχαίουμε το ταμείο αυτό με άλλα ταμεία και αυτό δεν είναι σωστό, ιδιαίτερα το κοινωνικό. Δεν θα πρέπει να υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στα δύο αυτά ταμεία. Ευχαριστώ, Μάριαν. Thank you, Thank you, Madam President. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για ε, την ε, έκθεσή της. Ε, θα ήθελα όμως να προτείνω μια αλλαγή. Στην παράγραφο 6 αναφέρεται την άδεια της χρήσης του Ταμείου ως ένα μέσο επέμβασης στην απώλεια θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω συμφωνιών που έχουν συναυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν το θεωρώ δίκαιο ούτε για τους εργαζόμενους ούτε για, τους, ούτε για τις επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν πέσει θύματα των εμπορικών διαφωνιών δεν είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έλαβαν τις λάθος επιχειρη... Ε, αποφάσεις, όμως φέρουν το βάρος, ε, είναι αυτοί που πραγματικά χάνουν. Για παράδειγμα, πάρτε το ρωσικό εμπάργο. Ε, πα, ε, το τομέα τροφίμων έχει επηρεαστεί σοβαρά από το συγκεκριμένο εμπάρκο. Οι συνέπειες έχουν ω αποτέλεσμα μικρές ομάδες ε, να ε, σηκώνουν το βάρος, το συνολικό βάρος της διαμάχης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωση και Ρωσία. Θέσεις εργασίας έχουν χαθεί, όμως το εμπάρκο επηρεάζει διάφορες περιοχές, ε, θέσεις εργασίας, ε, τομείς εργασίας και κράτη-μέλη. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει ε, να προσθεθεί ένα σημείο το οποίο θα υποστηρίξει επιχειρήσεις οι οποίες επηρεάζονται από εμπορικές διαφωνίες και υποστηρίζω εντόνως τη συγκεκριμένη πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε μήπως η Κομισιόν ε, να προσθέσει κάτι πριν δώσω το λόγο ε, στην κυρία Χάρκιν. Θα είμαι πάρα πολύ ε, σύντομη. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι η αναφορά της κυρίας Χάρκιν είναι πάρα πολύ χρήσιμη και αναγνωρίζει τις αλλαγές που έχουν γίνει με βάση την νομοθεσία κατά την περίοδο 2007-2013. Συμφωνούμε ότι το Ταμείο έχει έναν ε, ρόλο ως ένα εργαλείο αλληλεγγύης λόγω των αλλογών στην αγορά. Όμως θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το Κοινωνικό Ταμείο έχει, ένα, έχει μια συγκεκριμένη αποστολή, δηλαδή να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις οι οποίες περιμένουν ε, τις ε, αλλαγές. Ε, δεν περιμένουμε λοιπόν το Ταμείο Προσαρμογής να το κάνει αυτό, διότι για αυτό υπάρχει το Κοινωνικό Ταμείο συμφωνώ ε, ότι ε, ότι πάντοτε το 100% ε, των ανθρώπων που θα, στους οποίους θα απευθυνθούμε δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιτεύξιμο. Θα ήθελα να σας πω ότι η Κομισιόν ζητάει συνεχώς περισσότερες πληροφορίες από τα κράτη-μέλη και αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, θα πρέπει μέσα σε έξι μήνες από την ολοκλήρωση της επέμβασης να παραδώσουν μια αναφορά και εδώ θα ήθελα να αναφερώ, αναφερθώ σε κάποια κράτη-μέλη τα οποία διστάζουν ε, να κάνουν αρκετά διαφανή τη διαδικασία αιτήσεων. Θα ήθελα να συγχαρώ λοιπόν τα κράτη-μέλη τα οποία το έχουν κάνει αυτό ε, δημόσια διαθέσιμο δύο φορές το χρόνο θα ε, πρότεινα να υπάρχει ε, μια συνάντηση ε, με τους εθνικούς συντονιστές και θα ζητούμε όταν τα κράτη-μέλη ετοιμάζουν μια αίτηση να χρησιμοποιούν τα μέσα που ορίζονται από το άρθρο 4.2 Μέχρι στιγμής ακούσαμε ότι μπορεί, μπορεί να υπάρχουν διοικητικές ελλείψεις όσον αφορά ε, την αίτηση για κάποιες επιχειρήσεις, ιδιαίτερως ε, τις μικρομεσές, όμως εμείς δεν σταματούμε να υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη ε, και σε αυτές τις συναντήσεις λοιπόν τα κράτη-μέλη παρουσιάζουν τις υποθέσεις τους και ε, υπάρχει δυνατότητα λοιπόν ε, για τους εκπροσώπους των κρατών μελών να λάβουν πληροφοριοδότηση σχετικά με, τις, ε, με τα σχέδια τα οποία έχουν επιτυχημένως χρηματοδοτηθεί. Το Κοινοβούλιο επίσης συμμετέχει στην αξιολόγηση των υποθέσεων. Σας συγχαίρουμε επίσης για τον περιορισμό των χρονοδιαγραμμάτων. και μέχρι στιγμής μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα και να δικαιολογήσουμε ε, αποδείξεις με βάση τις υποθέσεις που έχουν, έχουν χρηματοδοτηθεί. Έχουμε πάνω από 100 υποθέσεις και μπορούμε να αναλύσουμε μονάχα αυτές οι αποδείξεις λοιπόν που έχουμε είναι περιορισμένες, δεν έχουμε ακούσει ακόμα για χρήματα τα οποία εξαφανίζονται από τα ταμεία λόγω της φύσης της εφαρμογής και η Κομισιόν πραγματοποιεί ελέγχους, δεν κάνουμε μονάχα έναν άλογχο, αυτό είναι ξεκάθαρο και όταν γίνονται έλεγχοι τότε αυτό γίνεται σε συμφωνία με, τους, ε, με τις εθνικές υπηρεσίες και ε, ε, επίσης ε, οι δικοί μας ελεγκτές αποδέχονται τα δεδομένα των εθνικών υπηρεσιών. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για αυτήν την αναφορά από την κυρία Χάρκιν. Συμφωνούμε με τα περισσότερα σημεία που αναφέρονται και πιστεύουμε λοιπόν ότι σίγουρα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, όμως τώρα απαιτείται περισσότερη εμπειρία και δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χάρκιν. Μια και έχω δύο λεπτά, δεν θα μιλήσω πολύ. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία δυσυστήθηκαν. Σημειώσα όσα υπόθηκαν από του συναδέλφου. Σύντομα θα θέλω να αναφερθώ σε ζητήματα που δεν είχαμε θίξει σε προηγούμενε συζητήσει. Ένα από αυτά το φέρατε εσείς, Πρόεδρε, ένα πλαίσιο για την αλλαγή και την αναδιάρθρωση, που να το συζητήσουμε διμερώς. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το ενσωματώσω, αλλά βεβαίως πολύ ευχαριστώ να το συζητήσουμε. Αρκετοί συνάδελφοι είπαν ότι δεν είναι γνωστό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να προβάλλουμε την ενημέρωση. Βεβαίως και οι εργαζόμενοι, όπως και οι πολιτικοί δεν το γνωρίζουν. θα χρησιμοποιήσω, εάν χρησιμοποιήσω μόνο μία λέξη σε σχέση με το Ταμείο, θα χρησιμοποιήσω αυτή που έφερε η Μαρία Ρενά, προσθετικότητα δηλαδή, γιατί αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση, δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Και επίσης, πολλοί έθιξαν, το έχουμε ζητήσει βέβαια και στο παρελθόν, αλλά πολλοί υπογράμμισαν ότι χρειάζεται μια πιο προνοητική δράση σε σχέση με τους εργαζόμενου από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μαθαίνω από την Επιτροπή ότι οι τελικέ εκθέσει ορισμένων κρατών δεν ήταν απαραίτητα διαθέσιμε. Νομίζω ότι εμεί ω Κοινοβούλιο θέλουμε να δούμε τι εκθέσει αυτέ. Θέλουμε διαφάνεια. Για τον κύριο Κρίστιανσεν. Η παράγραφο 6 για να σας ε, παραπέμψω στην προηγούμενη πρόταση του τρέχοντος κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρότεινε λοιπόν εκεί η Επιτροπή να περιλαμβάνονται και οι γεωργείς. Αυτό δεν είχε συμφωνήσει στο Κοινοβούλιο, γιατί αυτό είχε θεωρηθεί ως φίλος εκείς για μια συμφωνία Μερκασούρ που θα έχει συνέπειες σε διάφορους τομείς της γεωργίας. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε και είναι διαφορετικό το επιχείρημα από ό,τι είχαμε συστήσει τότε. Αλλά δεν ήθελα κανένας ε, επίτροπος εμπορίου τρέχον, τρέχουσα ή προηγούμενος να μου πει ότι με 150 εκατομμύρια το χρόνο μπορούμε να λύσουμε προβλήματα των ε, συνεπειών των προτάσεων αυτών. Βέβαια, εσείς μιλάτε για κάτι διαφορετικό, μιλάτε για εμπορικές διαμάχες, που θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Αν λοιπόν δεν έχω αναφερθεί σε παρατηρήσει των συναδέλφων, όλων των συναδέλφων, παρακαλώ μην νομίζετε ότι σα αγνώρισα, απλώ ε, για να μπορέσουμε να τελειώσουμε εγκαίρω, συνόψα στα απαραίτητα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο. Βεβαίω βλέπουμε ότι υπάρχει μια πλήρη και ολοκληρωμένη στράτευση από πλευρά σα για το θέμα του Ταμείου Παγκοσμιοποίηση. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 25 Απριλίου σύντομα δηλαδή. Εξέταση 24 Μαΐου, ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 15-16 Ιουνίου, Ολομέλεια κατά τις προβλέψεις μετά τις θερινές διακοπές, ίσως το Σεπτέμβριο. Και με αυτά νομίζω εξατλήσαμε την ημέρηση διαταξή για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 9 το πρωί και ξεκινούμε εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας της Κορέας.